η έκθεση της κυρίας ε, Τόματσης ε, παράκτη αλία μικρής κλίμακας στις περιοχές που εξαρτώνται από την ε, αλία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, Επίτροπε κύριε Βέλα, αγαπητοί συνάδελφοι. Το σύνθημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενωμένη στη διαφορετικότητα, πολυμορφία, έχει υπάρξει γενικό. Η πολιτική όμως ε, ε, αυτή ήταν ε, μέχρι τώρα ενιαία και όχι, δεν είχε έλαβε υπόψη τις διαφορές. Κάποια θέματα που αφορούν στη μικρή κλίμακα παράκτια ηλία είναι παράδειγμα. Τα κράτη-μέλη αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο και ως εκ τούτου έχουμε ένα νομοθετικό πλαίσιο που περιορίζει την ανάπτυξη των αλληλευτικών κοινοτήτων και στην Νότια και στην Βόρεια Ευρώπη. Το πρώτο βήμα για την ανάπτυξη του νέου πλαισίου θα πρέπει να καθορίσει την ε, μικρή κλίμακα παράκτια ε, αλληλεία και την παραδοσιακή αλληλεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, λαμβάνοντα υπόψη τι ιδιωτερότητε των διαφόρων αλληλευτικών περιοχών. Ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει υπόψη τα διάφορα ενδεικτικά κριτήρια για όπως το μέγεθος των, ε, πλοίων, τα ελληνικά εργαλεία, την επιλεκτικότητα των τεχνικών, το, τη διάρκεια των αλλιευτικών ταξιδιών αλλά και διάφορα άλλα τοπικά χαρακτηριστικά όπως την επίπτωση της ε, αλίας αυτή, στην ευημερία της τοπικής κοινότητας. Θα πρέπει να, ληφθεί, να επανεξεταστεί η σημασία της ε, μικρής κλίμακας ε, παράκτης αλίας στις νησιωτικές περιοχές οι οποίες εξαρτώνται για την επιβίωσή τους. Η διάκριση αυτή θα είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με τη νέα πρωτοβουλία για τα νησιά Πού που ε, παίρνει υπόψη τους λύσεις στο πρόβλημα της οικονομικής και δημογραφικής ε, ε, παρακμής των νησιών. Πρέπει επίσης να περιοριστούν οι αρνητικές επιπτώσεις της γραφειοκρατίας και γι' αυτό ζητάμε από την Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να εξασφαλίσει ότι η μικρής κλίμακας παράκτη αλία θα χρηματοδοτηθεί επαρκώς από το EFF Επίσης, η παραδοσιακή αλία είναι σημαντικό κομμάτι της ιστορικής και παραδοσιακής κληρονομιάς ε, των παρακτήων περιοχών και κοινοτήτων και προωθείται, μπορεί να προωθήσει τον τουρισμό. Θέλουμε στο, η Αλία να συμπεριληφθεί στον τομέα των τεχνών και πολιτισμού. Αλλά για να εξασφαλίσουμε το βιώσιμο μέλλον των νησιωτικών κοινοτήτων, η έκθεσή μας είναι υπέρ της διαφοροποίησης της Αλίας με την ανάπτυξη συμπληρωματικών δραστηριοτήτων, της επένδυσης σε σκάφη και εξοπλισμό, την ανάπτυξη της κατάρτισης και της καινοτομίας. Άρα οι βασικοί στόχοι πρέπει να είναι ε, να προωθηθούν ε, πρωτοβουλίες που θα είναι βιώσιμες μέσα οικονομικά και περιβαλλοντικά. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο με την εμπλοκή όλων των ενδιαφερομένων πλευρών, ερευνητικών κέντρων, πανεπιστημίων, ε, των τεχνολογικών κέντρων, τοπικών και περιφερειακών Ινστιτούτων. Ζητούμε λοιπόν ε, από την Επιτροπή να δώσει τις απαραίτητες συνθήκες που θα μπορέσει να να προωθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση και να δώσει καλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Εν κατακλείδη θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι συμμετείχαν στην σύνταξη της έκθεσης αυτής. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τους κοιόδης εισηγητές και τα μέλη της Επιτροπής Αλίας, των οποίων η πρόταση και η συμμετοχή στις συζητήσεις βοήθησαν στην δημιουργία μιας επικοδομητικής και θετικής ατμόσφαιρας. Ως εισηγήτρια όμως θα ήθελα να ευχαριστήσω τους, τους Κροάτες ειδικού και αλληλείς, οποίοι με την ευκαιρία αυτή προσέφεραν την τεχνογνωσία και την εμπειρία τους για τη διαμόρφωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Μια ε, ανοιχτή και ειλικρινή επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκομένων και των πολιτικών ξεκινά μια νέα διαδικασία και μας δίνει την ελπίδα ότι μαζί με τους Ευρωπαίους πολίτες θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε αυτά που πρέπει να βελτιωθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Πολύ και προχωράμε στη δικασία Catch the Eye. Πρώτος είναι ο Φρανσίσκο Χωσέ Μιανμόν. Για ένα λεπτό. Ε, Εμείς χαιρετίζουμε αυτή την έκκληση γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η παραγγελία. Είναι το 66% του στόχου του δικού μας και στην ε, Γαλλική. Είναι το 85% των σκαφών. Δηλαδή έχουμε πάνω από 3.800 ε, σκάφη. Και πάρα πολύ πρόσφατα η Επιτροπή Αλληλείας έκανε αποστολή εκεί και είδε τι γίνεται με την παραδοσιακή αλληλεία και τι γίνεται με τα σκάφη εκεί, με τις επιχειρήσεις που είναι οικογενειακές, τους τρόπους ε, αλληλείας, τους συγκεκριμένου, και είδαμε ότι βοηθά το περιβάλλον αυτή η αλληλεία, καταναλώνεται και λιγότερο ε, πετρέλαιο και καύσιμο. Οπότε βλέπουμε ότι αυτό το Ταμείο της ε, Αελίας αναλαμβάνει κάποιες πρωτοβουλίες για την ανταγωνιστικότητα του παραδοσιακής σαλία στην Γαλλικία εφαρμόζεται αυτό το πρόγραμμα, τρέχει αυτό το πρόγραμμα για τον παραδοσιακό αλληλευτικό στόλο και υπάρχουν διάφορα ε, μέτρα για απασχόληση ε, για την υποδοχή της μίας γενιάς από την άλλη στην απασχόληση και επίσης και να υπάρχει περισσότερη αποτελεσματικότητα από τα σκάφη. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Σάντος είναι επόμενος ομιλητής για ένα λεπτό. senhor comissário parece me importante reconhecer que há neste relatório uma defesa muito interessante das pescas nas zonas mais remotas ou seja nas zonas ultraperiféricas da Europa. De facto, nos Açores, de onde... Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι αυτή η έκθεση φροντίζει για τα συμφέροντα των εξόχως αποκέντρων περιοχών και έτσι μπορούμε να προστατεύσουμε τα μικρότερα σκάφη και αυτή η προσέγγιση έχει επιστημονική τεκμηρίωση. Νομίζουμε ότι έτσι θα δοθούν ευκαιρίες οικονομικής ε, προόδου, θα προστατευτεί επίσης και το περιβάλλον. Η βιοποικιλότητα, αλλά και υπάρχουν πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της εκπαίδευσης των ε, αλλία. Συμφωνούμε με αυτά που λέει η έκθεση και νομίζουμε ότι το ταμείο αυτό, το EMFF, μπορεί να καλύψει τα συστήματα που χρησιμοποιούνται ε, και μπορεί το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θερασκελίας να χρησιμεύσει εμπειρία και για άλλους τομείς. Ευχαριστώ πολύ. Επειδή βρισκόμαστε πολύ καλά, πάμε πολύ καλά με το χρόνο μας, θα συμπεριλάβω όλους τους ομιλητέ που θέλουν πάρουν το λόγο. Ο κ. Μαριά είναι ο επόμενο ομιλητή. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε η παράκτη αλληλεία αποτελεί μια κοινωνικά βιώσιμη μορφή αλληλείας η οποία σύμφωνα με την κοινή αλλιευτική πολιτική μπορεί να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα και την επιχειρηματικότητα στον αλλιευτικό τομέα. ωστόσο σε πολλά κράτη μέλη της ένωσης οι παράκτιες και νησιωτικές περιοχές αντιμετωπίζουν σημαντική οικονομική ύφεση που έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του πληθυσμού και την φυγή των κατοίκων. επιπλέον σε χώρες όπως η ελλάδα που πλήττεται από τα μέτρα της λιτότητας και του μνημονίου οι αλλοίς βιώνουν τις συνέπειες του αγροτικού μνημονίου της τρόικας με αποτέλεσμα την οικονομική ύφεση η οποία είναι πολύ πιο έντονη. είναι επομένως αναγκαίο η ευρωπαϊκή ένωση να λάβει άμεσα μέτρα ώστε να ανασυγκροτηθεί ο πρωτογενής τομέας να δοθεί έμφαση στη γαλάζια οικονομία να ενισχυθεί η απασχόληση στις παράκτιες και νησιωτικές περιοχές και να αυξηθεί η χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής ένωσης στον αλλιευτικό τομέα ενώ σε σχέση με την ελλάδα θα πρέπει επιτέλους να μπει φραγμός στην φορομπηχτική λαιλασία και στο αντιασφαλιστικό ρεσάλτο στα πενιχρά εισοδήματα των αλλιέων. ευχαριστώ. Επόμενη ομιλήτρια είναι η κυρία Μπιλμπάου Παραντίκα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Πιτρό, η κοινή αλληλευτική πολιτική χρειάζεται ε, μια περιχαράγωση του τομέα πράκτη πράκτης γιατί είναι πάρα πολύ κρίσιμο αυτός ο τομέα, η δραστηριότητα αυτή για τον κόσμο και για πρώτη και αυτή την ε, πολιτιστική παράδοση, την ελληνική παράδοση ε, δεν, δεν ωφελεί να ασχολούμαστε με το μέγεθο μόνο και την ισχύ του κινητήρα των σκαφών. Θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με την αελία μικρή κλίμακα και από την άλλη μεριά με την παραδοσιακή αελία των παρακτήων περιοχών. Ε, θα πρέπει να σκεφτούμε το πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί η αιλία e, ακόμα και για ε, ψυχαγωγία ε, για τον τουρισμό γιατί όλα αυτά είναι πολιτική κληρονομιά της Ευρώπης και θα πρέπει να σκεφτούμε επομένως το πώς θα καλύψουμε τους μέλλοντες υπάλληλου του σήματος του ευρωπαϊκού τουρισμού. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Φερέρα έχει το λόγο για ένα senhora Η μεταρρύθμιση της ε, αλληλευτικής πολιτικής δεν έλυσε τα προβλήματα της ε, παράκτειας αλίας. Το αντίθετο, πολλά από τα προβλήματα παροξύνθηκαν, άρα θα πρέπει με την παρούσα ευκαιρία να ε, δούμε το πώς θα μπορέσουμε να επεξεργαστούμε ένα κοινοτικό πρόγραμμα και για αυτήν την μορφή αλίας. Τέτοια θα πρέπει να είναι η προσέγγιση μας, έτσι να είναι η διαχείριση. Θα πρέπει να προστατευτούμε προς την κοινοτομία να καλύψουμε όλο τον αλληλευτικό στόλο, να φροντίσουμε και τα εισοδήματα των άλλων, ε, Να εξασφαλίσουμε επίσης και δίκαιες τιμές του προϊόντος να δούμε πώς θα προστατεύσουμε τις ε, παρακτικές ε, κοινότητες, πώς θα υπάρχει κατά προτεραιότητα πρόσβαση στους πόρους. Επομένως θα πρέπει να αναλυθεί δράση, να θεσπιστούν μέτρα, περισσότερα μέτρα από όσα έχουν γίνει μέχρι σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ ο κύριος Σταφόσκη, για ένα λεπτό. Ε, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να συγχαρώ την κυρία Τόμασιτς για την εξαιρετική αυτή έκθεση που βοηθά στην βελτίωση της θέσης των ε, αλλιέων η νέα αυτή προσπάθεια που ξεκίνησε τον, Ιούνιο, τον Ιανουάριο του 2014 θα πρέπει να βοηθήσει τους ε, αλληλείς. Η βελτίωση της ζωής στις παράξεις περιοχές δεν θα είναι δυνατή μέχρι ότου ε, υπάρξει ο μεσογειακός κανονισμός ο οποίος ασχολείται με τα παραδοσιακά λευτικά μέσα και τεχνικές στη Μεσόγειο. Η η, κατάσταση, η παρούσα κατάσταση έχει ε, οδηγήσει σε, ε, ε, δημογραφικό μαρασμό των νησιών και θα πρέπει να οριστεί η μικρή κλίμακα παράκτια αλία και η παράκτια αλία σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες των περιοχών και όχι μόνο σε σχέση με το μέγεθος και την δυναμικότητα των σκαφών. Και γι' αυτό πιστεύω ότι ο κανονισμός δεν είναι παρικής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Όλοι συμφωνούμε ότι είναι αναγκαίο να κάνουμε μια προσπάθεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να προστατεύσουμε την παράκτη αλληλεία. Μιλούμε για έναν τρόπο ζωή που πρέπει να διατηρήσουμε αλλά και για μια κοινωνική και οικονομική δραστηριότητα που θα πρέπει να είναι βιώσιμη εάν λάβουμε τι αναγκαίε αποφάσει, ειδικού κανόνε για ειδικού τύπου αλληλεία. Και αυτό είναι σημαντικό ιδιαίτερα για ορισμένε ε, περιφέρειες όπως οι από κέντρες ε, ε, περιοχές που χρειάζονται ειδική προστασία για να αγγιθούμε την επιβίωση των αλλιέων που χρησιμοποιούν παραδοσιακές πρακτικές αλλίες. Η παράκτια αλλία είναι θεμελιώδης για την οικονομική ανάπτυξη αυτών των περιφερειών λόγω των γεωγραφικών τους χαρακτηριστικών και τη μεγάλη τους απομάκρυνσης από, τα, από την υπηρετική χώρα. Θα πρέπει λοιπόν να προωθήσουμε καινοτομίε που μπορούν να εγγυηθούν την χρηματοδότηση αυτών των παραδοσιακών αλλιευτικών σκαφών. Επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Νικολά Καπούτο για ένα λεπτό. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Η Επιτροπή θα πρέπει να προσπαθήσει να υποστηρίξει κάποιο προγράμματα καινοτομία και θα πρέπει να μπορέσουμε να αναπτύξουμε αυτή την αλλήλεια. Και αυτό θα πρέπει να λάβει προτεραιότητα και έτσι να μπορέσουμε να σώσουμε θέσεις εργασίας και επίσης να προστατεύσουμε την παραδοσιακή αλληλεία και όλες τις σχετικές γαστρονομικές δραστηριότητε. Θα πρέπει επομένως να υπάρξει ποικιλία στους τρόπους ε, αλληλεία, να προστατεύσουμε μόνο τις τοπικές κοινότητες, ε, τους διάβλους ε, του τοπικής διανομής του αλλιεύματος και επίσης το, θα πρέπει τα κράτη-μέλη προοδευτικά να επιτύχουν αύξηση των ποσοστώσεων για την παραδοσιακή αλία γιατί και από κοινή πλευρά είναι πάρα πολύ σημαντική ευκαιρία. πρέπει να γίνει βιώσιμη και θα πρέπει να υπάρξει χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Ελίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ και τώρα ο κύριος Γιάκοφτσιτς έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε πολιτική για την Αλία ε, μοιάζει να έχει επενεθεί από κάποιο γραφειοκράτη, από κάποιους γραφειοκράτες στις ε, Βρυξέλλες. Η έκθεση αυτή είναι ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα καρπός μακρών διαπραγματεύσεων και σκληρής προσπάθειας. Γι' αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία εισηγήτρια και να εκφράσω την υποστήριξή μου προς αυτήν και θα ήθελα η μικρή κλίμακα παράκτη αλία να έχει την θέση που της αξίζει εντός της ευρωπαϊκής πολιτικής. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την επιβίωση πολλών αλλίων στα νησιά καθώς και για την προώθηση του τουρισμού και για την γαστρονομία των νησιών και των παράκτιων περιοχών. Θα ήθελα να εκφράσω τη στεναρή μου υποστήριξη για αυτή την έκθεση και θα ε, υποστηρίξω την έκθεση αυτή στην Κροατία και στις άλλες ε, περιφερειακές ε, περιοχές της Ευρώπης. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Τόμασικ για την έκθεσή της και την πρότασή της να, μεταρρυθμιστούν, να μεταρρυθμιστεί ο κανονισμός για τη Μεσόγειο όσον αφορά τη, τη μικρής κλίμακας παράκτη αλία που είναι ιδιαίτερα σημαντική για τις ε, νησιωτικές και παράκτιες περιοχές της ε, Κροατίας. Γι' αυτό θα πρέπει να προσθεθεί, να συμπεριληφθεί μάλλον στον ε, κατάλογο της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κροατίας οι παράκτιες ε, κοινότητες πάσχουν ήδη από αφέμαξη του πληθυσμού. Η μικρή κλίμακας ε, ε, βιοτεχνική αλία ε, σε αυτά μια παράδοση πολλών αιώνων και είναι αναπόσπαστο στοιχείο της κροτικής ε, πολιτιστικής ταυτότητας. Γι' αυτό χρειάζεται μια περιφερειακή προσέγγιση όσον αφορά την ε, διαχείριση των αποθεμάτων και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας όλα τις βιολογικές και οικολογικές και γεωγραφικές ιδιαιτερότητες εάν θέλουμε να αναχαιτήσουμε τα αρνητικά αποτελέσματα της ε, αλληλευτικής πολιτικής μέχρι τώρα. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Γελέρα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ την κυρία Τόμαση γιατί πραγματικά έκανε μια εξαιρετική δουλειά. Ε, έλαβε υπόψη της όλες τις ε, προτάσεις και νομίζω ότι γέννη η έκθεσή της είναι πολύ επαρκής. Θα ήθελα να τονίσω κύριε Πίτροπε, ότι όλοι οι συνάδελφοι αναφέρθηκαν ότι είναι αναγκαίος ένας νέος ορισμός της ε, παράκτιας ε, ε, βιοτεχνικής μικρής κλίμακας αλίας. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει ένας νέος παρκέστερος ορισμός. Βεβαίως ε, είναι αναγκαία και μια υποστήριξη. Μέχρι στιγμής ε, κάτι τέτοιο δεν, δεν έχει γίνει. Επίσης θα πρέπει να δημιουργηθεί, ε, να προωθηθεί ένας κλάδος τουρισμού στον οποίο να μπορεί να συμμετάσχει αυτός ο τομέας και να μην, αυτός ο κλάδος και να μην αποκλείεται από αυτόν. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριο Κούν είναι τελευταίο ομιλητή στη διαδικασία Κατσουδιά για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Αξιότιμη κύριε Βέλα. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό σε έναν βασικό κανονισμό να συμπεριλάβουμε την ε, μικρής κλίμακας ε, παράκτια βιοτεχνική αλία και να μεριμνήσουμε για τα αναγκαία χρηματοδοτικά εργαλεία προκειμένου να υποστηρίξουμε ε, αυτού του τύπου αλεία γιατί ένα μεγάλο ποσοστό ε, συμπεριλαμβάνεται σε αυτή την μορφή αλίας. Γι' αυτό είναι σημαντικό εδώ και το στοιχείο της ε, περιφερειοποίησης. Θα ήθελα λοιπόν ο κ. Βέλλας να δώσει μια ελευθερία στις χώρες μέλη, δηλαδή να μην μπει one size ε, fits all, αλλά να μερμνήσει για πολλαπλά διαχειριστικά σχέδια, τα οποία να είναι επαρκώς ε, προσαρμοσμένα στις διάφορες ε, περιοχές. Για την περιοχή της Βαλτικής, ευτυχώς, έχουμε εκπονήσει το διαχειριστικό πρόγραμμα το οποίο λαμβάνει υπόψη του τα, τις κοινωνικές ε, ενισχύσεις που πρέπει να δίνονται εγκαίρως και διάφορα άλλα στοιχεία ούτω ώστε να μπορέσουν να γίνουν και οι κατάλληλες επενδύσεις στο πλαίσιο του σχεδίου Juncker και να πάμε προς την ορθή κατεύθυνση. Ευχαριστούμε ε, και πάλι και τώρα ο κ. Ε, Βέλλας έχει εξ ονόματος της Επιτροπής το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αγαπητά μέλη. Χαιρετίζω την ε, έκθεση Δίας Πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την καινοτομία και διαφοροποίηση παράκτης αλληλείας μικρής κλίμακας περιοχές που εξαρτώνται από την αλλία και θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια την κυρία Τόμασιτς για την εξαιρετική έκθεση. Το, Ευρωπα... το Ευρωπαϊκό Ταμείο ε, Θάλασσας και Αλληλείας υποστηρίζει την κοινή αλληλευτική πολιτική για το διάστημα 2014-2020. Και αυτό ήταν το αποτέλεσμα έντονων διαπραγματεύσεων μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Χάρη στο Ταμείο, τα κράτη-μέλη μπορούν και κατά πάσα πιθανότητα θα πραγματοποιήσουν τα περισσότερα από όσα προτείνονται και ζητούνται στην έκθεση. Το Ταμείο προσφέρει ε, ε, ενίσχυση 80% σε όλους όσοι ασχολούνται με την μικρή κλίμακα ε, παράκτη αλληλεία, όπως ας πούμε το ξεκίνημα νέων αλλιέων, η ασφάλεια και η υγιεινή συνεργασία, κατάρτιση, διαβιομάθηση, θέματα εμπορίας και επεξεργασίας και κοινοτομίας. Όμως τα κράτη-μέλη έχουν την ευθύνη να, για να αποφασίσουν με βάση τα διάφορα επιχειρησιακά προγράμματα ε, που έχουν ε, εγκριθεί μέχρι το 2015 πώς θα επιλέξουν τις προτεραιότητες και θα προσφέρουν συγκεκριμένη υποστήριξη. Ε, είναι πολύ αποκαλυπτικά τα στοιχεία, διότι είναι περίπου τα 3 τέταρτα, δηλαδή το 75% των ε, ενεργών αλληλευτικών σκαφών. Είναι μόνο 12% της ε, αξίας των ε, ελευμάτων και 16% ε, του συνολικού ΑΕΠ, αλλά ε, μεγάλο ποσοστό, 36% ε, του, του αντίστοιχου πλήρους απασχόλησης που σημαίνει ότι ένα μεγάλο μέρος των θέσεων εργασίας είναι μερικής απασχόλησης. Αυτό σημαίνει ότι η αλληλεία δεν είναι η μοναδική ή ούτε καν η βασική βασική πηγή εισοδήματο για πολλού από του παράκτιου αλληλεί και τι οικογένειέ του. Και παρά τα αυτά, ε, είναι γεγονό ότι πολλά από τα αλληλευτικά σκάφη είναι θεμελιώδου σημασία για την βιωσιμότητα των ε, παρακτίων κοινοτήτων που εξαρτώνται από αυτά. Συμφωνώ απόλυτα με την άποψη αυτή. Είναι όμω γεγονό ότι η βιομηχανική αλληλεία η μεγάλη, ε, υπάρχει επίση στι παράκτιε περιοχέ και εκεί. Ε, ε, έχουμε τις μεγαλύτερες, ε, τα, μεγαλύτερα ποσά και ε, την απόδοση. Άρα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Επιπλέον το, το απλό ποσοστό ότι έχουμε 36 περίπου αποθέματα στον Ατλαντικό σε MSY μπορούν δείχνει ότι μπορούμε να έχουμε και εδώ βιώσιμη αλληλεία με κοινωνικά ωφέλη. Με βάση όλα αυτά πρέπει να στηρίξουμε τον αλληλευτικό στόλο και να αποφύγουμε τη δημιουργία μιας ασύμετρης αλληλευτικής πολιτικής παρότι αναγνωρίζουμε και την μεγάλη σημασία της μικρής κλίμακας παράκτια αλληλεία. Όσον αφορά τις απαιτήσει για τον έλεγχο θα πρέπει να πω ότι ε, υπάρχουν προτιμησιακοί όροι στήριξης από το για την παρακτιαλία, για την εγκατάσταση ε, ε, ε, εξοπλισμού στα πλοία. Και όσον αφορά τον, την αναθεώρηση του κανονισμού για τον έλεγχο, πρέπει να προσέξουμε, να αποφύγουμε, να προκληθεί μια ε, κίνδυνος εξάντλησης των, των αλληλευτικών στις περιοχές όπου ε, ε, αλλιεύουν οι παράκτη αλληλείς και όπου υπάρχουν προτιμησιακές ε, ρυθμίσεις από τα κράτη-μέλη. Θα μπορούσε να η παράκτια αλία να δημιουργήσει πρόβλημα στην περιοχή των 12 ναυτικών μιλίων, ιδίως σε περιοχές όπου υπάρχει μεγάλη πίεση για, τις, ε, για τα ελεγχόμενα και μη ελεγχόμενα ε, αποθέματα. Αυτό πιστεύω ότι αυτό θα, έχει, θα βλάψει και την οικονομική βιωσιμότητα και το περιβάλλον. Όσον αφορά τον ορισμό της, ε, μικρής, του μικρού μεγέθους ε, παράκτης αλίας, ο κανονισμός 314 ε, καλύπτει σκάφη λιγότερο, μικρότερο των 12 μέτρων που δεν χρησιμοποιούν εξοπλισμό θέμα που συζητήθηκε έντονα στον τριμερή διάλογο για τον κανονισμό και αναφέρεται στο σημείο 1 της έκθεσης όπου προτείνεται, αναλύεται και συζητείται αλλά δεν, δεν κατέστη δυνατόν να ε, καταλήξουμε σε απόφαση για τον ορισμό. διότι θα υπήρχε ο κίνδυνος δημιουργίας ανισοτήτων. Εν κατακλείδη, όλοι οι στόλοι συμπεριλαμβανομένου και του αλλιευτικού στόλου μικρής παράκτιας αλλίας είναι σε θεμελιώδους σημασίας για τις παράκτιες περιοχές και πρέπει να φροντίσουμε να πετύχουμε την ε, περιβαλλοντική οικονομική και οικονομική και κοινωνική βιωσιμότητα των παράκτων περιοχών. Υπάρχει μεγάλη στήριξη προς αυτή την κατεύθυνση από, από την κοινή γνώμη και η χαλάρωση των απαιτήσεων για έλεγχο και η ανάπτυξη της αύξησης της ζώνης των 12 ναυτικών μιλίων θα απειλήσουν την αντοχή αυτών των κοινοτήτων. Δεν έχω αμφιβολία ότι οι συνομοθέτες θα επανέλθουν στο θέμα αυτό στο πλαίσιο του, του σχεδιαζόμενης αναθεώρησης του κανονισμού αυτού. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε. Εδώ ολοκληρώνεται η συζήτηση και η ψηφορία θα διεξαχθεί αύριο. Και τώρα